Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση που είναι η πρώτη μας συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές. Θα θυμάστε ότι πριν από έξι εβδομάδες, ε, στις 19 Ιουλίου, είχαμε συνεδρίαση με τον Επίτροπο Χόγκαν, που μας ενημέρωσε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας για την κατάσταση στο γαλακτοκομικό τομέα και το πακέτο του γάλακτος, όπως ε, έχει γίνει γνωστό το πακέτο των μέτρων. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω όλους στην πρώτη μας αυτή τη συνεδρίαση μετά το καλοκαίρι, τους ευρωβουλευτές, ε, τους υπαλλήλους, τη γραμματεία, τους διερμηνείς, Ελπίζω όλοι να αναπαυθήκατε και να γυρίσετε ακμαίοι για το δύσκολο έργο που σας περιμένει. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε την αγαστή μας συνεργασία και σήμερα και στη συνέχεια. Έχετε λάβει το σχέδιο μερίσης διάταξης. Και μάλιστα το πρωί θα έχουμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης μια κυκλισμένα των θυρών συνεδρίαση των συντονιστών. Καταρχήν να, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Δεν υπευλήθησαν σχόλια για την ημερήσια διάταξη, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνεται όπως σας έχει υποβληθεί. Μάλιστα να μεταδίδεται και από το διαδίκτυο και έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες με εξαίρεση τεστονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά. Ε, θα ήθελα να κρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 25ης Μαΐου και 20ης-21ης Ιουνίου. Θα ακολουθήσουμε την γνωστή διαδικασία και να περάσουμε στο σημείο 4. Ε, θα τα εξετάσουμε, θα τα ψηφίσουμε από κοινού τα σημεία 4 και 5 γιατί αφορούν και τα δύο το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δημοσιονομικό έτος 2017. Όλα τα τμήματα. Η συγητής της γνωμοδότησής μας είναι ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάρ έχει πλούσια πείρα γιατί πολλές φορές έχει ασχοληθεί με τα δημοσιονομικά ζητήματα. Οπότε θα ψηφίσουμε για το σχέδιο της γνωμοδότησης και τις ε, δημοσιονομικές, τις ε, τροπολογίες των προπολογισμό. Ξέρετε ότι η αιτήσια διαδικασία για τον προπολογισμό διαιρείται σε πολλές φάσεις και μάλιστα στις 14 Ιουλίου ε, ψηφίσαμε τη, την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Γιάρ κατέπτυσε τη σχετική γνωμοδότηση και συζητήθηκε στην 14η Ιουλίου και μάλιστα μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 62 τροπολογίες για τη γνωμοδότηση. Ο εισηγητής, σε συνεργασία με τους και οδησηγητές, συνέταξε μία συμβαστική πρόταση που καλύπτει όλες αυτές τις ε, τροπολογίες. Σε αυτό το πρώτο της ψηφοφορίας θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή μας, τον κύριο Γιάρ, για να μας κάνει την εισαγωγή για την ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης πρώτα. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας σε όλους τους συναδέλφους. Ξανά ήρθαμε στις Βεξέλλες μετά το καλοκαίρι και αρχίζουμε με τα νυφάλια θέματα, προϋπολογισμό και γεωργικά. Ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι η πολιτική που μεταφεράζεται σε αριθμούς. Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά εδώ τους και ηγητές συναδέλφους γιατί είχαμε πρόβλημα και αυτή είναι μια κριτική που πρέπει να διαβιβάσω εγώ και επιθυμώ να διαβιβάσω στον Πρόεδρο της Επιτροπής μας. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αριθμητικά ήρθαν πολύ αργά λόγω του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Και ακόμα πιο αργά τα αριθμητικά στοιχεία ε, του Συμβουλίου. Την τερκούας ε, εβδομάδα ε, δημοσιεύτηκαν αυτά εκλογικής περιφέρειας. Και χθε το βράδυ έπρεπε εκτάκτω να κάνουμε συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και ευχαριστώ πάρα πολύ του συναδέλφου που μπόρεσαν και ήρθαν. Αλλά κανονικά θα πρέπει να το πούμε και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι δεν είναι σοβαρή αυτή η ε, εργασία. Για να δουλεύουμε σοβαρά θα πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο και την ευκαιρία να ε, διαβουλεύεται. Και επειδή εγώ είμαι εκφύσεω αισιόδοξο, Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα τα ε, κάνουμε καλύτερα. Ε, ποια είναι τώρα εδώ η βασική ιδέα ε, και η κεντρική ιδέα στις διαβουλεύσεις. Καταρχήν, σήμερα ψηφίζουμε. Θα δείξει η ψηφοφορία πώς θα συμπεριφερθούμε. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τις περικοπές του Συμβουλίου και να επανέλθουμε στο σχέδιο του προπολογισμού που καθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να το πω και λίγο σαρκαστικά, χειρότερα δεν γίνεται. Έχουμε συνεννοηθεί με τις πολιτικές ομάδες να προβλέψουμε χρήματα επιπλέον για έκτακτες περιστάσεις, θεομηνίες και απρόβλεπτα έτσι, συμβάντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Επίσης, εκφράσαμε πάλι τη λύπη μας για τις περικοπές. Θα γίνει ένας ανταγωνισμός ιδεών εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε καλά δεν θα γίνουν αυτές οι περικοπές στην πράξη. Αυτά είναι θεωρητικά γιατί ε, πάντα υπάρχουν κάποιες ε, αρχικές δυσκολίες αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην χάσουμε τα χρήματα αυτά επαγίως τα επόμενα χρόνια. Ε, και καλό και κακό νέο έχω στα πιλωτικά προγράμματα. Χαίρομαι ε, για ε, τις περιφέρειες που προβλέπονται εδώ πολλά πιλωτικά προγράμματα, αλλά τι να πρωτοδιαλέξουμε. Έχουμε βάλει συν σε όσα προγράμματα έχουν βαθμολογία Α και Β. Θα τα ξαναδεί η Επιτροπή Προπολογισμών αυτό. Ευχαριστώ πάντω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν ε, για τα πιλωτικά προγράμματα. Ε, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε την προσπάθειά μας. Καλύτερα να έχουμε πολλά προγράμματα και να επιλέγουμε παρά να παραμελούμε τις ε, περιφέρειές μας. Από πλευρά γεωργικής πολιτική. τα του προπολογισμού είναι γνωστά. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ούτε τίποτα εθεροβάμονες είμαστε και ονειροπόλοι, αλλά στην ενδιάμεση αναθεώρηση και το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό μας έταξαν κάποια κονδύλια. Αυτά θέλουμε να τα δούμε να ε, αφιερώνονται στη συγκεκριμένη πολιτική. Δεν μειώθηκαν τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία επειδή έχουμε προβλήματα κι αλλού. Το αντίθετο θα έλεγα. Άρα αυτό ε, θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να το λέμε και στους αγρότες και να δεσμευόμαστε γιατί περιμένουν να το ακούσουν από εμάς. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν όλους τους όλες για τη συνεργασία και ε, τη χτεσινοβραδινή συνεδρίαση που έγινε τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Δεν ζητά κανείς το λόγο για απορίες ή ερωτήσεις προς τον εισηγητή, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Νομίζω ότι όλοι έχετε φέρει τις ε, κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές, σας το είχα πεθυμίσει άλλωστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Εγκρίνεται. 15 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 19. Τροπολογία 19. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. 21. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 22. Ο εισηγητής μας παρακαλώ. Εδώ ε, υπάρχει μια προφορική τροπολογία, μια διόρθωση μεταφραστική. Ήθελε ο συντάκτης ε, να αρνηθεί την περικοπή στον προϋπολογισμό και μάθαμε ότι η σωστή λέξη στα αγγλικά είναι reject και όχι refuse επειδή ήθελε να ε, απορριφθεί, δεν ξέρω στη μητρική του αλλά στα αγγλικά λέγεται αυτό reject για την απόρριψη όχι refuse. Αυτό είναι γλωσσικό απλώς για να διορθωθεί και να γίνει ε, σωστή η τροπολογία και να εκφραστεί και αυτό που επιθυμούσε ο συντάκτης. Ευχαριστώ. Αναφέρεται άλλωστε και στον κατάλογο ψηφοφορίας αυτή η αντικατάσταση. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογίας 22. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά απορρίπτεται 27 υπέρ κατά απορρίπτεται ...28 για το ίδιο θέμα με την 22 οπότε δεν χρειάζεται να δώσουμε τις ειδικές εξηγήσεις. Ποιος είναι υπέρ του 28 εγκρίνεται, ευχαριστώ Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 29. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. ανεπαίσθητη η διαφορά, δύσκολο να τη δούμε με το μάτι, οπότε σωστά το ελέγξαμε ηλεκτρονικά. 30 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα για την 31, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 32, 33 και 34 από κοινού. Δεν βλέπω αντίρρηση. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Α, όχι. Διαφωνείτε. Πρώτα την 32 τότε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά απορρίπτεται και αυτή 34 υπέρ κατά απορρίπτεται 35 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 35 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 40 υπέρ, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 42 και 50 ταυτόσημες μαζί. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 43. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 46, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Α. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά της συμβαστικής τροπολογίας Α. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, υπάρχει ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ας επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Επανάληψη της ψηφοφορίας της ηλεκτρονικής. Ας αφαιρεθεί μία ψήφος από τους σοσιαλιστές. Ένας παρακαλώ μη ψηφίζει. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία Α. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 48 υπέρ κατά απορρίπτεται 49 υπέρ εγκρίνεται 51 υπέρ κατά κατά τη γνώμη μου απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πενήντα τέσσερα της κυρίας Σένερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, αλλά οριακά. 56 το κύριο Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 57. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 59 υπέρ, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 61 υπέρ, εγκρίνεται. 62 υπέρ, εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδότησης ε, μετά την έγκριση και των τροπολογιών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα των ψηφοφοριών, ψηφοφορία των συγκεκριμένων δημοσιονομικών τροπολογιών με τα ποσά, Μας εξήγησε τα θέματα ο εισηγητής μας. Τέλη Ιουλίου πήραμε τα, τις προτάσεις με τα συγκεκριμένα ποσά, 20 Ιουλίου. Και ήταν πολύ ε, βραχίες οι προθεσμίες λάβαμε υπόψη κυρίως ε, τις εκτιμήσεις για τις προτάσεις του Συμβουλίου. Ε, τα πιλωτικά σχέδια εντάσσονται στην εντολή της, ε, της ψηφοφορίας για τις δημοσιονομικές τροπολογίες και όπως ξέρετε γίνονται απευθείας οι τροπολογίες αυτές στην Επιτροπή Προπολογισμού μετά την προκατακτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκανε μια ταξινόμηση και αξιολόγηση των πιλωτικών σχεδίων και στην πράξη ε, γίνονται, δεκτές, ε, γίνονται δεκτά τα πιλωτικά σχέδια που έχουν λάβει βαθμολογία Α και Β κυρίως. Μόνο αυτές, αυτά τα σχέδια έχουν μεγάλη πιθανότητα έγκρισης. Μόνο για τα σχέδια που έχουν λάβει Α και Β υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα υπόλοιπα πολιτικά πιλωτικά σχέδια δεν έχουν μάλλον πιθανότητα να εγκριθούν. Τέτοια τα πρακτική ακολουθούν και άλλες επιτροπές, δηλαδή ψηφίζονται οι προτάσεις των πιλωτικών σχεδίων που έλαβαν υψηλή βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά τα Α και Β. Και μάλιστα ε, υπευλήθησαν και κάποιες προτάσεις για πιλωτικά σχέδια στην Επιτροπή Γεωργίας που δεν αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τις ψηφίσουμε και αυτές μαζί με τις υπόλοιπες προτάσεις πιλωτικών σχεδίων που έχουν λάβει υψηλή βαθμολογία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι άσχετα με την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της, θα έχετε την ευκαιρία να καταθέσετε εκ νέου τα πιλωτικά σχέδια και απευθείας στην Επιτροπή Προϋπολογιζών μέχρι την 5η 1η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να προσθέσει ο εισηγητής μας. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία των δημοσιονομικών τροπολογιών. Τροπολογία πρώτη, 5766, πρώτο τμήμα. που αφορά το ύψος των ποσών. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε, τις 5766, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της 5766 που αφορά το κείμενο. Ποιο είναι υπέρ του δεύτερου τμήματο της τροπολογία αυτής. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 57-50. Ποιος είναι υπέρ. 57-50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. Τροπολογία 57-55. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-59. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-54. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-63. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-52. Υπέρ εγκρίνεται. 57 77, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 57-86, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 57-56, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 57-78, ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται 57-73 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 57-60 ποιος είναι υπέρ να την μαζί με την 57-83 γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ εγκρίνονται τροπολογία 57-81 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 57-79 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος. Θέλετε. Ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 5775. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Μόη το ζήτησε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5775. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορια Απορρίπτεται. Τροπολογία 5776. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 57-80 υπέρ κατά απορρίπτεται. 57-84 υπέρ κατά απορρίπτεται. 57-87 υπέρ κατά απορρίπτεται. 57-68 Ποιος είναι υπέρ. Νομίζω ομόφωνα εγκρίνεται. 57, 80, α, συγγνώμη, καταπίπτει αυτή, 57-89, πάμε στην 57-90. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 57-91, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 57-92. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-64. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-69. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-93. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-53. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 57-94. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-60. 70 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57-57. Υπέρ. Εγκρίνεται. 57-71 υπέρ κατά απορρίπτεται 57-61 υπέρ εγκρίνεται 57-95 υπέρ κατά απορρίπτεται 57-72 υπέρ μαζί με την 5796 ε, από κοινό υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 57-58 υπέρ, εγκρίνεται. 57-65 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 57-62 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 57-51. Υπέρ. Εγκρίνεται. 58 Νέο πιλωτικό σχέδιο. Ψηφίζουμε για νέο πιλωτικό σχέδιο. 58-00. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 58-01. σχέδιο παρόμοιο με τα 58-13. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 5802, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. 5803 υπέρ κατά απορρίπτεται. 5804 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 5805 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 5805. Άρχεται η ψηφοφορία. απορρίπτεται. Κατά τη γνώμη μου. Αλλά για θέμα αρχής, όντως απορρίπτεται. 58.06 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 58.07 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 58.08 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5809 υπέρ κατά απορρίπτεται 5810 υπέρ κατά απορρίπτεται πιλωτικό σχέδιο 5813 αποσύρεται με θετική σύσταση αλλά καλύπτεται με καλύτερη διατύπωση από την τροπολογία 5801 που ούτως ή άλλως έχει εγκριθεί. Περνάμε στην τροπολογία 5767 του κυρίου Μπέλντερ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5798. Σρέιρ και Μαγκίνες. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Και τελευταία τροπολογία, 57-97. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίσαμε και τις τροπολογίες των προπολογισμό. Στις 11 Οκτωβρίου θα εγκρίνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών το ψήφισμα για τον προϋπολογισμό. Στις, στις 26 ε, Δεκάτου θα εγκριθεί η θέση του Κοινοβουλίου στην ανάγνωση. 28 Οκτωβρίου ξεκινάει η διαδικασία των 21 ημερών για την περίοδο της συνδιαλλαγής που ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε την 1η Δεκεμβρίου την έκβαση της συνδιαλλαγής. Οπότε μπορείτε να, βάλτε στη τσέπη σας πια τις ηλεκτρονικές κάρτες. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, δεν χρειάζονται. Περνάμε στο σημείο 6, την επένδυση στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της ε, συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Αξιολόγηση με βάση το άρθρο 16, παράγραφος 3 του Κανονισμού Περί Κοινών Διατάξεων. Η συγκήτριά μας που συνέταξε και τη γνωμοδότηση είναι η κυρία Νταντσίλα. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εμείς απλώς γνωμοδότηση καταρτίζουμε. Στις 15 Μαρτίου αποφασίστηκε η σύνταξη της γνωμοδότησης ε, επί της έκθεσης πρωτοβουλίας ε, μη νομοθετικού χαρακτήρα ε, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Επαναλαμβάνω, μη νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπότε θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Τάντσιλα, που ήδη στις 24 Μαΐου μας παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησης. Σήμερα η κυρία Δαντσίλα θα μας παρουσιάσει και το σχέδιο, μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψε, το σχέδιο της γνωμοδότησής της. Μετά την παρουσία της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Νταντσίλα, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα διαστατικά και επενδυτικά ταμεία και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι βασικοί μηχανισμοί ε, για τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Αλλά και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ε, πώς θα επενδύσουμε στην οικονομία γιατί ε, είναι δύσκολη καιρή και χαλεπική για την οικονομία και για την πολιτική. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και προσπάθησα να εστιάσω στα προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου ε, για ε, το ταμείο αυτό, το ΦΕΝΤΕΡ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης που έρχεται να τονώσει και να αναζωογονήσει τη γεωργική ανάπτυξη για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, προηγούμενα προγράμματα ήταν πιο περίπλοκα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουν απλουστευτεί και έχουν γίνει και πιο ευέλικτα έτσι ώστε να απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιφέρειας. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο ρυθμός των στρατηγικών στόχων έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την καινοτομία, το περιβάλλον και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που είναι τρεις εγκάρσιοι οριζόντιοι στόχοι. στόχοι. αυτα αυτά ορισμένα κράτη-μέλη και ορισμένες περιφέρειες δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως και να εκμεταλλευτούν την αυξημένη κατά τα άλλα ευελιξία των ταμείων. Για ποιο λόγο διότι η έλεγχη ήταν πιο πυκνή και η περιπλοκότητα παρέμενε, παρόλο που είχε απλουστευτεί το πρόγραμμα. Θα πρέπει να βγάλουμε λοιπόν τα συμπεράσματά μας από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, από τη λειτουργία του Ταμείου και τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι ώστε στο μέλλον να προλαμβάνουμε τυχόν καθυστερήσεις. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ποια ήταν η δυνατότητα απορρόφησης ε, των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ευελιξία αυτή που παρέχουν οι δύο πυλώνες με αύξηση της εθνικής συμμετοχής. Ονομαστικά μέχρι σήμερα ήταν με, ε, μείωση αυτή που παρατηρήθηκε ως προς το ποσό ε, σε σχέση με την περίοδο 2007-2014, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η ευελιξία και η δυνατότητα μεγαλύτερης εθνικής συμμετοχής, υπήρξε τελικά κάποια αύξηση. Μικρή μεν, αλλά αύξηση. Ε, κατά τη σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής διαπίστωσα ότι ε, στα ε, επιχειρησιακά προγράμματα και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης γίνονται δράσεις μόνο όταν συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς. Όχι μόνο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και διάφοροι από την κοινωνία των πολιτών. Έτσι και μόνο έτσι επιτυχάνουν τα προγράμματα αυτά σε τοπικό επίπεδο και είναι και σωστή και αποτελεσματική η διαχείριση των πόρων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω με χαρά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Νταντσίλα. στη συζήτηση. Ο κύριος Λαζό ζήτησε πρώτα στο λόγο, παρακαλώ. Oui, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά τα ταμεία ε, αυτά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, οι ε, επενδύσεις, το λέτε κι εσείς μόνοι σας, οι λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες έτσι θα μπορέσουν ε, να φτάσουν στις πιο ανεπτυγμένες. Δηλαδή, ε, συνειδητά διοργανώνεται μία, έναν ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα με την διερμηνία στα αγγλικά. Okay. Εντάξει τώρα. Συνεχίσω. Ο κύριος Λουαζό. Λέω λοιπόν ότι οργανώνεται πλέον ε, ένας ανταγωνισμός μεταξύ ε, των κρατών μελών. Για το 2014-2016 ο πίνακας 1 είναι πάρα πολύ εύγλωτος. Ε, ευνοείται τις ανατολικές χώρες όπως το είχατε ξανακάνει για τα σιτηρά και διακυβεύονται καλλιέργειες χωρών όπως η Γαλλία, δυτικών χωρών. Εδώ έχουμε χρήματα των ε, Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, υπέρ των μεταναστών, υπέρ των προσφυγών, των προσφύγων ε, και μετά από όσα έγιναν στη Γερμανία με τον ανταγωνισμό που πληρώνονται λιγότερο οι πρόσφυγες έχουμε και έναν ανταγωνισμό εις βάρος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και οι μεγάλοι όμιλοι που πιέζουν, απασχολούν πρόσφυγες και μετανάστες με χαμηλότερους μισθούς εις βάρος ε, των πολιτών. Και έχετε και βίκορους από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα αιτήματα. Τι γίνεται με τους Γάλλους αγρότες. Θα πρέπει να ετοιμαστείτε να τρέχετε πάρα πολύ γρήγορα όταν θα σας κυνηγήσουν, γιατί τους συναντάω συχνά και ξέρω τις διαθέσεις και τις προθέσεις τους δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κακή απέναντί μας και τόσο απειλητική η Γεωργία τη Χριστή να τα βάλουμε στα πόδια. Παρακαλώ κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τη συντάκτρια γνωμοδότης κυρία Τάντσιλα για την έκθεσή της που είναι μια καλή αφετηρία και μπορούμε από εκεί και πέρα να εργαστούμε και εμείς και να κάνουμε και κάποιες προτάσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τίτλος της έκθεσης, δηλαδή η βελτιστοποίηση της συμβολής των ταμείων για την ε, ανάπτυξη και της, την απασχόληση. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Το λέει και στη γνωμοδότησή της η Στο σημείο 2 λέει ότι τα ε, επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία είναι βασικά εργαλεία και εκ των όνου Εγώ θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Η προσθετικότητα αυτών των πόρων και των ταμείων ε, είναι εκ των όνου έτσι ώστε να αναπτυχθεί η υπεθρός και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Προσθετικότητα. Καμιά φορά, το θυμόμαστε όλοι, πώς ξεκίνησε η συζήτηση για το σχέδιο Juncker. Απέκλειε την ύπεθρο και εμείς χρειάστηκε ειδικά να το διεκδικήσουμε αυτό ε, για να συμπεριληφθεί. Άρα λοιπόν η προσθετικότητα των ταμείων των πόρων, δηλαδή να αθρίζονται και στην ε, σύνταξη μια τέτοια γνωμοδότηση, εμεί ω Επιτροπή Γεωργία θα πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις και στόχους ε, ε, για τους νέους και τις γυναίκες της υπαίθρου. Αλλιώς δεν πρόκειται να αναπτυχθούν ούτε θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν. Αυτά τα δύο ήθελα να θέσω και φυσικά θα κάνω και τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Βιωρίκα ε, Νταντσίλα για τη γνωμοδότησή της και την ανάλυση της. Είναι πολύ εύστοχη και οξυδερκής και συμφωνώ μαζί της για την αποτελεσματικότητα της δράσης ε, στην απορρόφηση των ταμείων. Θα πρέπει αυτά όλα να γίνονται πολύ κοντά ε, στους αποδέκτες. Η επικορικότητα είναι η λέξη κλειδί και το έχουμε δει διαχρονικά. Όσο είμαστε πιο κοντά ε, σε εκείνους που διαχειρίζονται ε, αυτά τα προγράμματα, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε. Γιατί όταν γίνεται εκ του μακρόθεν η διαχείριση δεν βοηθάει και είναι ατελέσφορη. Μιλήσαμε και για το ποσό. Εντάξει, κάποια στιγμή, πώς να το πω, αν βρούμε περισσότερα λεφτά, καλώ. Και εδώ έρχομαι και στην προηγούμενη συζήτηση για το προπολογισμό του 2017. Τόσο το καλύτερο αν έχουμε περισσότερα χρήματα, αλλά τώρα έχουμε δυσκολίε. Και υπάρχει ένα θέμα ουσίας, πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια και ποιος ε, δικαιούται και νομιμοποιείται ε, και αν νομιμοποιείται αυτή η πολιτική στα μάτια των πολιτών. Το θέμα δεν είναι μόνο το ποσό, αν θέλουμε να συγκλίνουμε, που είναι και βασικός στόχος και υποχρέωσή μας, ε, αυτό είναι το ένα. Αλλά και το δεύτερο είναι ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση των προγραμμάτων. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να διατηρηθεί η ζωή στην Ήπεθρο και μάλιστα στις πιο δύσκολες περιοχές, θα πρέπει να πιάνουν περισσότερο τόπο τα κονδύλια αυτά, να είναι πιο έξυπνη η διαχείριση για να παραμένει ζωντανή η Ήπεθρος και σήμερα, κυρίως και αύριο. Άρα, θα κάνω και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να σκεφτούμε και τη μελλοντική ε, προγραμματική περίοδο της κοινή γεωργικής πολιτικής για το πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά τα διαστατικά ταμεία για τους πόρους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλκάρσελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρώτο θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ την κυρία Τανθήλα για την εξαιρετική ε, δουλειά της. Εδώ πρόκειται για ένα θέμα που έχει τεράστια σημασία. Δεδομένης και της κρίσης που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τη Γεωργία. Άρα τα διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιούμε τους ε, στόχους ε, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι ως προς τις προσαρμογές στη κλιματική αλλαγή, τα ενεργειακά, τα θέματα εκπαίδευσης κλπ. Αλλά στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της στόχιας απέχουμε από τους στόχους μας. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και ποιο τον αμφισβητεί. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να δοθεί και μία όθηση στην γεωργική αγροτική οικονομία στην Ήπεθρο. Ο ανταγωνισμός, όμως η ανταγωνιστικότητα των ε, επιχειρήσεων στην Ήπεθρο είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώ ο δεύτερο πυλώνας κοινή γεωργική πολιτική με την πάροδο του χρόνου έχει αποδυναμωθεί και ο πρώτος πυλώνας επίσης δεν έχει ενισχυθεί. Και βεβαίω η μεταφορά των πόρων από, το δεύτερο, από τον πρώτο συγγνώμη, στο δεύτερο πυλώνα δεν είναι λύση για να αναπτυχθεί η πεθρός Ούτε είναι καλή λύση να τα βγάζουμε από τη μια τσέπη για να τα βάζουμε στην άλλη. Έχουμε αυτό το αιώνιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, είναι πάρα πολύ απαραίτητο να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση που στραγγαλίζει ε, την κοινή γεωργική πολιτική. Αλλά δεν συμφωνώ με την υπεραισιοδοξία της ως προς τη μεταφορά πιστώσεων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Συνεπώ θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε τη σημασία ε, των ταμείων αυτών για την καταπολέμηση της φτώχειας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, με νέες τεχνολογίες, με έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα της ανεργίας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο, όπως λέει και η συγγήτρια, να Εκκινούν πιο γρήγορα τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου στην αρχή της κάθε προγραμματικής περίοδου. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα διότι χρονίζει και βαραίνει ε, την πολιτική αυτή εδώ και χρόνια. Επίσης χρειάζονται κατευθύνες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε ο αγροδιατροφικός τομέας να δει ότι υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μαζί ε, και σε συνδυασμό με το νέο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Τρει παρατηρήσει έχω να κάνω. Να ευχαριστήσω καταρχά την εισηγήστρια για την έκθεση. Ίσως έχουμε εκεί κάποιο χώρο να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Από πολιτική πλευράς για μένα είναι σημαντικό τα προγράμματα για την Επίτρο να διοικούνται, να την κάνουν διαχείριση από την Επιτροπή Άγκρη. Είναι σημαντικό δηλαδή από πλευράς ε, πολιτικής ε, αγροτικής να ε, παρακολουθούμε και την Ήπεθρο. Και υπάρχουν φυσικά και αρμοδιότητες και σε άλλες επιτροπέ, όπω η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και φυσικά είναι σημαντικό το θέμα αυτό γιατί σε πολλέ περιπτώσει ε, μα ρωτάνε τι κάνουμε στην Επιτροπή Αρτική Ανάπτυξη και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι εμεί θα πρέπει να παρακολουθούμε τα θέματα που αφορούν την Ήπεθρο. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημείο 10. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε λοιπόν και στην Ήπεθρο σωστά προγράμματα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των τοπικών παραγόντων και αυτοί θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι, να τολμούν να παρουσιάσουν προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ακόμα και να ενισχύσουμε το σημείο 10. Στο μεγαλύτερο πρόβλημα στο σημείο 8. Μιλάτε για over-regulation, για υπερβολική ρύθμιση. Ε, Ευτυχώ που το αναφέρετε, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτή τη ρημάδα την απογραφή κρυοποιητήση. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί υπάρχει έλλειμμα σε συγκεκριμένο τομέα. Ποια προβλήματα υπάρχουν δηλαδή για τη μείωση της γραφειοκρατίας και θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι περιφερειακές ε, αρχές και θα έπρεπε ενδεχομένω και με την ε, Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί φυσικά πάντα χρειάζονται έλεγχοι και πάντα πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσον υπάρχει διαφθορά, απάτη, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση μάλλον περιβάλλουμε. Και έτσι έχουμε τους αγρότες αφενός, τους γεωργούς, οι οποίοι λίγο πολύ έχουν συνηθίσει κάθε χρόνο να πολεμούν και να αγωνίζονται με τις ευρωπαϊκές ε, κατευθυντήριε γραμμέ, αλλά έχουμε και κάποιου ε, που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά στη ζωή του. Ε, για παράδειγμα, μια εταιρεία η οποία υποβάλλει μια ε, αίτηση για ένα project, για ένα έργο. Και αυτοί λοιπόν οι φορέί οι οποίοι για μία φορά μόνο συμμετέχουν χάνονται λίγο στη γραφειοκρατία και κάνουν λάθη. Εννοείται ότι κάνουν λάθη και αναγκάζονται να επιστρέψουν χρήματα. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν κάτι καλό και τελικά μπλέκουν. Και έτσι όλο και πιο πολλές, ε, ε, όλο και πιο πολλά παράπονα λαμβάνουμε και ενστάσεις και από τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες πλέον δεν είναι σε θέση να τα επεξέλθουν. Λόγω του όγκου της γραφειοκρατίας. Δεν καταφέρνουν να εφαρμόσουν όλα αυτά και αυτό προφανώς είναι επιβλαβές για τις ε, εργασίες μας. Άρα, να το τονίσουμε το σημείο 8 και να το τονίσουμε και παραπάνω από ό,τι τονίζεται. Αν δεν υπάρξει μείωση τη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, το στόχο μα. Να κινηθεί κάτι επιτέλου από οικονομική άποψη στην Ήπεθρο. Και θα πρέπει τα προγράμματα να είναι διαφανή και για αυτού που τα χρησιμοποιούν. Αν δεν έχουν μια αλφα επισκόπηση τη κατάσταση, θα είναι αντιπαραγωγικά και θα καταλήξουμε σε μια υπερβολική διαδικασία γραφειοκρατίας και ελέγχου. Στο σημείο 8 λοιπόν το τονίζω ιδιαίτερα. Το τονίζω μάλιστα γιατί ξέρω ότι έχει εντελώς αντίθετη ε, νότροπια και πορεία η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Εγώ θέλω να είναι ξεκάθαρα τα προγράμματα. Εντάξει, να μην υπάρχει δυνατότητα απάτης και διαφθοράς, δεν λέω, αλλά να είμαστε και σε θέση να επιτρέπουμε και ένα σφάλμα όπου δεν υπάρχει τουλάχιστον ε, δυνατότητα μεγάλης ε, απάτης ε, και μεγάλης ζημίας. Ιδάλλω θα καταλήξουμε να έχουμε ωραία προγράμματα στη θεωρία, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται στην πράξη. Και επίσης να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά την Ήπετρο, μας ενδιαφέρουν οι, μικροί, οι μικροί φορείς όχι μεγάλες ε, επιχειρήσεις των εκατομμυρίων. Γιατί αυτές οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις έχουν μια ολόκληρη ομάδα, έχουν μια ολόκληρη νομική υπηρεσία με δεκάδες δικηγόρους. Ε, οπότε αν τυχόν υπάρξει ευρωπαϊκός έλεγχος, έλεγχος από ευρωπαϊκής πλευράς, ε, τους παραπέμπουν αυτόματα στο νομικό τμήμα. Εμείς όμως θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για το μικρό φορέα, για το μικρό αγρότη. Πώς θα μπορεί αυτός να διαχειριστεί τα προγράμματα και να μην τιμωρηθεί επειδή έβαλε ένα λάθος κόμμα κάπου ή έκανε ένα μικρό σφάλμα κάπου. Και σας καλώ λοιπόν να αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Σήμερα παρά ήσασταν το κύριε Γιάρ. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Κυρία Σρέερ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά που μόλις είπε ο συνάδελφος Πετεργιάρ ήταν ακριβώς αυτά που ήθελα να πω και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά να σας ζητήσω το εξή. Το τελευταίο καιρό άκουσα το τι είπε ο συνάδελφος Μαλίστερο για το θέμα αυτό. Κοιτώντα λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία μετά το 2018, το 2020 θα αντιμετωπίσουμε λιτότητα στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της υπέτρου, δύο πράγματα έχω να πω. Καταρχάς αυτό που είπε ο κύριος Γιάρ και το λένε και άλλοι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ειδικού για θέματα ε, επιδοτήσεων και έτσι οι πολυεθνικές ε, μαζεύουν όλα τα χρήματα, όλες τις επιδοτήσεις ε, και αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία και οι Ολλανδοί αγρότε πολλέ σε πολλέ περιπτώσει στρέφονται στη Γερμανία, ενώ οι μεγάλες, οι μικρέ ε, οικογενειακέ επιχειρήσει δεν ξέρουν πώ να τα βγάλουν πέρα και τι να κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Αυτό σχετίζεται και με το ταμείο το επενδυτικό του Juncker, αλλά και πρέπει να σας πω ότι είμαι υπέρ του τη διαχείριση του κλίματο, τη βιοπικιλότητα κτλ. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η διατήρηση τη υπαίθρου για το πράσινο, για του αγρότε κτλ. Στο μέλλον λοιπόν, Πού θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε χρήματα για αυτού του ανθρώπου οι οποίοι φροντίζουν ακριβώ αυτού του στόχου μα μετά το 2018, μετά το 2020, γιατί ω Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσουμε μια αλφαξιοπιστία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολλούς βουλευτές και πολλοί έχουν απόψεις από αυτού. Άλλωστε, αυτό είναι και ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε απόψει, τοποθετήσει. Αλλά σε πολλέ περιπτώσει η προετοιμασία των εγγράφων παίρνει πάρα πολύ χρόνο και τελικά χάνεται η ουσία ενδεχομένω του θέματο. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νταντσίλα, εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ σορροπημένη η δουλειά που έκανε την έκθεση αυτή. Και αυτό πρέπει να πω ότι παρουσιάζει ένα ενίο και ομοιόμορφο σύνολο, το οποίο εστιάζεται στα πιο σημαντικά στοιχεία. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ΚΑΠ και το πώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία χρηματοδότηση ε, τη ανάπτυξη τη υπέτρου. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί η γραφειοκρατία και να μπει πιο έντονο το στοιχείο τη ευελιξία. Ίσως να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο της καινοτομίας της τεχνολογικής αλλαγής που κινείται με ταχύς ρυθμούς, ιδιαίτερα στην ε, Ήπετρο. Και αυτό ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα και για την βιωσιμότητα του κλάδου αυτού στην Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή λοιπόν, Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει λίγο πιο δραστήριο ρόλο στα ζητήματα αυτά, να διαβιβάσει στους αγρότες το μήνυμα ότι έχουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένε δυνατότητε. Και το θέμα λοιπόν τη γραφειοκρατία μα απασχολεί ιδιαίτερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νταντσίλα για τι προτάσει που κατέθεσε. Θα καταθέσω κάποιε τροπολογίε, αλλά θα είναι ίσονο σημασία και μάλλον θα ήθελα με αυτέ να τονίσω κάποια ζητήματα για να αλλάξω την ουσία. Ευχαριστώ κύριε Σάγκελο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτά που συζητάμε λοιπόν είναι η περιπλοκές που προκύπτουν από τα επενδυτικά προγράμματα στα θέματα τα αγροτικά. Ο κύριο Γιάρ λοιπόν πήρε το λόγο, αλλά να τονίσω ότι είναι ένα γερμανό βουλευτέ. και αν αγωνίζονται και δεν τα βγάζουν πέρα οι Γερμανοί αγρότε, που ξέρουμε ότι αποτελούν την κινητήριο ε, δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και αυτοί λοιπόν θα βρίσκουν σκούρα έχουμε πρόβλημα. Το πρόσφατο δημοψήφισμα ε, για τον Brexit ε, μα εξέπληξε το πώς οι αγρότες ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης της ε, Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, θα μπορούσατε να κλείσετε το μικρόφωνο αυτό. Ο κύριος Ντε μιλάει και με ενοχλεί. Μιλούσα λοιπόν για την, ε, το δημοψήφισμα για τον Brexit στη Βρετανία. Μα ξανάρχισαν να μιλάνε. Σας ευχαριστώ. Πολλοί λοιπόν αγρότες ε, ψήφισαν υπέρ της εξόδου. Και ένας λόγος, ένας από τους λόγους είναι το πόσο περίπλοκο είναι ε, να τα βγάλει κανείς πέρα μέσα στο δέταλο των εγγράφων που χρειάζεται για να πάρει κανείς μια χρηματοδότηση. Και ξέρει, ε, ξέρει ο κόσμος ότι ε, χάνουμε χρήματα από τον πρώτο πυλώνα που πάνε στον δεύτερο πυλώνο και ότι άλλοι τελικά υποφελούνται. Αυτά α, θεωρούν, αυτά βλέπουν ε, οι Βρετανοί αγρότες. Τι γίνεται λοιπόν με τους Βρετανούς φορολογούμενους. Ε, οι φορολογούμενοι ξέρουν ότι δίνουμε διπλά από αυτά που παίρνουν οι αγρότες και προφανώς ε, χρειάζεται και θέλουν να υπάρχει σωστή, σωστός α, έλεγχος της χρηματοδότησης. Αλλά τελικά τα χρήματα αυτά πού θα καταλήξουν σε κάθε, κατά πάσα πιθανότητα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μεταφέρουμε χρήματα από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα και να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια αυτά για τους μετανάστες στη Γερμανία και σε άλλες χώρες από τις διάφορες χώρες της Βορείου Αφρική. Και θα ήθελα να σας προκαλέσω. Βγείτε και διαβεβαιώστε μου ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί δεν το είπα αυτό στην Επιτροπή πριν από κάποιες εβδομάδες ο Επίτροπος ε, δεν το αρνήθηκε κατηγορηματικά και νομίζω ότι προηγουμένως στην ψηφορία ήταν τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών λέξεων. Άρα, πείτε μου λοιπόν, κάντε σχόλια για το ότι τα κονδύλια από τον δεύτερο πυλώνα θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και την ε, συντήρηση των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο. Η παρουσία στην Ένωση και η συμμετοχή στην Ένωση δεν είναι μόνο ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού και αφαίρεση ε, η αξιοποίηση των κονδύλιων του προϋπολογισμού, αλλά και το ωφέλη της ενιαίας αγοράς, της κοινής αγοράς. Και ακόμη και χώρες που είναι περισσότερες συνεισφορείς έχουν καλύτερη ε, και πιο αναπτυγμένη δημοσιονομική υποδομή και αξιοποιούν καλύτερα τα ωφέλη της ε, κοινή αγοράς. Είναι αλληλένδετα αυτά τα θέματα. Και αναφέρεται συχνά ότι ακόμη και αν η συνεισφορά μερικών κρατών είναι μεγαλύτερη και τα ωφέλη είναι επίσης σημαντικότερα. Γιατί και είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την ανάλυση που έχει γίνει και πρόσφατα και δείχνουν ε, τα ωφέλη των ε, χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα από το ύψος της συνεισφοράς τους. Βέβαια, στο μέτρο που κάποιες ε, χώρες αναπτύσσονται, χάνουν το δικαίωμα για κάποια κονδύλια. Αλλά το καλύτερο είναι να μπορεί να, καθεί, να μπορεί να σταθεί μια χώρα στα πόδια της γιατί το ότι δεν είναι πια επιλέξιμη για συγκεκριμένα κονδύλια σημαίνει ότι μπορεί πια να τα βγάζει πέρα μόνη τη. Ε, και δείχνει ότι το αναπτυξιακό τη επίπεδο έχει βελτιωθεί. Ευχαριστώ και ε, συμπαθάτε με που έκανα αυτή τη σκέψη, αλλά νομίζω ότι ήταν καλή ευκαιρία. Κύριο Ροπέ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω... Πιστεύω ότι το σημερινό θέμα είναι από τα πιο σημαντικά που εξετάζουμε και αξίζει ενδελεχούς συζήτησης. Και φυσικά θα πρέπει να αξιοποιούμε σωστά τα κοινοτικά κονδύλια και να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας την μέχρι τώρα για να το επιτύχουμε, ώστε να πιάνουν τόπο τα κοινοτικά κονδύλια. Και ξέρουμε πιο είναι το οικονομικό, το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ποιο ήταν ε, και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα διάφορα κονδύλια, αλλά διαβεβαιότητα, τα διαρθρωτικά κονδύλια δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στην ε, Λιθουανία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά περισσότερο για τις υποδομές. Και οι επιχειρήσεις ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά τα αποτελέσματα ήταν μάλλον πενιχρά. Θα πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος, ε, να μάθουμε το μάθημά μας και να βοηθήσουμε αυτή τη φορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Και αν θέλουμε να μειωθούν οι ανισότητες και οι διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που μένουν πίσω να καλύψουν το έδαφος και να πλησιάσουν τις πιο αναπτυγμένες, ε, και να μην χρειάζονται οικογένειες ε, να ξενιτεύονται ή να ξενιτεύεται ο πατέρας για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του αναζητώντας δουλειά σε άλλη χώρα, θα πρέπει επιτέλους ε, να υιοθετήσουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και σε γεωργικά θέματα. Ήδη είχαμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από μια τέτοια προσπάθεια στη Λιθουανία. Και οι νέε θέσει απασχόληση δεν θα πρέπει ε, να δημιουργούνται ει βάρο των προηγούμενων. Σίγουρα θέλουμε νέε θέσει εργασία, αλλά να διαφυλάξουμε παράλληλα και τις ε, παλιέ θέσει εργασία και να μην τι καταστρέφουμε, να τι αναπτύσσουμε. Όλες αυτές ε, οι θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να δίνουν ελπίδα και προοπτική στον κόσμο και να μπορούν οι συμπολίτες μας ε, να προσβλέπουν σε έναν αξιοπρεπή μισθό και σε μια δίκαια αμοιβή για την εργασία τους. Επίσης θα πρέπει να διαφυλάξουμε όσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε. Γιατί αν δημιουργούμε τη μία θέση εργασίας και την επαύριο της καταστρέφουμε, δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο για να χρηματοδοτήσουμε και στο μέλλον τις θέσεις που δημιουργούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας για το έργο της. Και πριν ε, συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που είναι πολύ ενδιαφέρουσα για το πώς θα βελτιστοποιήσουμε και θα μεγιστοποιήσουμε τη συνεισφορά των διαρθρωτικών και παιδευτικών ταμείων που συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντική συζήτηση και θα συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή και στο έργο που γίνεται. Πρώτα απ' όλα όμως εγώ θα ήθελα να πω στην Επιτροπή μας ότι ένα από τα πρώτα σημεία που θα έπρεπε να εξετάσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα επενδυτικά ταμεία ω ε, μέσο εκβιασμού προ τα κράτη-μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μια τέτοια συμπεριφορά, γιατί πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί την Πορτογαλία και την Ισπανία με διακοπή των διαρθρωτικών και επενδυτικών κονδυλίων σε περίπτωση που δεν εκπληρώσουν ε, του στόχου ε, δημοσιονομικής προσαρμογής αυτός είναι εκβιασμός. Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η κρίση που βιώνουμε, η κρίση που μαστίζει του συμπολίτε μας και πώς επηρεάζει την απασχόληση, την ύπεθρο, και πόσο ενισχύει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφεύγει τέτοιου εκβιασμού. Θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα και το θάρρο να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παίζει με τα κρατημέλη, να μην τα απειλεί και να μην εκβιάζει του λαού τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, κυρία Σένερα. Ο κύριο Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με κάτι που είπε ο πρόεδρος απαντώντας στον βουλευτή Άγνιο για τα ωφέλη ε, της κοινή αγοράς, συμφωνώ και μου αρέσει και πάρα πολύ η ιδέα της κοινή αγοράς. Το πρόβλημα είναι ότι όταν παίρνει την κοινή αγορά και την τυλίγεις με μία σημαία και της βάζεις και ένα ύμνο και αφαιρείς κυριαρχία, δεν είναι κοινή αγορά, αλλά είναι ένα κράτο, πράγμα που εμεί δεν θέλουμε και δεν ήθελε ο λαό μα Έχουμε καταψηφίσει δύο φορέ τη συνδίκη τη Λισαβόνα και ελπίζω να ήταν αυτό μια αφύπνιση το Brexit και να ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του λαούς που δυστυχώ δεν συνέβη. Ε, καλό είναι λοιπόν που συζητούμε για το θέμα που μας απασχολεί και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω για τις δικές σας περιφέρειες, αλλά εκεί που ζω εγώ, πραγματικά η ύπεθρος ρημάζει, αιμορραγεί, φεύγει ο κόσμος, αποψηλώνεται γιατί τα χρήματα που θα έπρεπε να πάνε στην Ήπεθρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τελικά ε, πέφτουν στα χέρια γεωκτημόνων ε, και διαφόρων λεφτάδων που κυκλοφορούν με ιδιωτικά αεροπλάνα, τζετ και οι αγρότες αυτοκτονούν, γιατί στραγγαλίζονται, γιατί πραγματικά η ζωή τους είναι ένα μαρτύριο. 80% των ε, κονδυλίων ε, της γεωργικής πολιτικής και μετά το φύλλος εκεί της αναθεώρησης πηγαίνει στο 20% των πιο πλουσίων ε, γεωργών. Και μας λένε ότι παράγουν τόνους τροφίμων. Καθόλου τόνους, το 13% δεν παράγουν μόλις. Δεν θα πρέπει να επενδύουμε σε μεγαλογεωκτήμονες και τσιφλικάδες που κυκλοφορούν με ιδιωτικά τζέτ. Και δεν θα πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή ακούω εγώ απλώς ε, για ένα χρήσωμα της κατάστασης και πώς θέλει ο κύριος Χόγκαν ε, να τα ενισχύσει και κυρίως τον πρώτο πυλώνα. Και καθόλου δεν με εκπλήσει, γιατί αν το δείτε ιστορικά, υποφελείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε κάτι να απλουστεύσετε, απλουστεύστε το δεύτερο πυλώνα, γιατί είναι τέτοιο το χάος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας αγρότης που να έχει ε, χρόνο για να καλλιεργήσει ή για να ε, ε, δουλέψει την επιχείρησή του. Μόνο χαρτιά θα συμπληρώνει. Έχουμε μπει στο περιβάλλον, τους έχουμε κάνει τους αγρότες και πουρούς και τα λοιπά, αλλά αυτό που θα πρέπει να γίνει να πείσουμε τους αγρότες και να μας υποστηρίξουν και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τη γεωργία, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό όταν πάρα πολλά λεφτά δεν πηγαίνουν στην τσέπη των αγροτών και δεν μένουν και στην Ήπεθρο. Γιατί ένα πράγμα ξέρω να σας πω, ότι αυτός με το ιδιωτικό αεροσκάφος που κυκλοφορεί και ξοδεύει τα λεφτά του, δεν τα ξοδεύει στην Ήπεθρο, στην Ιρλανδία στο ίδιο κρεβάτι κοιμάται, σε ένα κρεβάτι κοιμάται και ένα γεύμα και ένα ύπνο τρώει τη μέρα. Δεν επενδύει τα χρήματα στην Ήπεθρο και θα πρέπει να πηγαίνουν στον τελικό αποδέχτη και όχι στους μεγάλο τσιφλικάδες αυτά τα λεφτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα σχόλιά σας και οι ερωτήσεις σας είναι πολύ εύστοχα και πολύ σημαντικά εν ώψη και τη ε, συζήτηση. Ε, και ελπίζω να τα σημείωσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Φεράν. Ευχαριστώ. Το ευρωπαϊκό πρότυπο των πατέρων ιδρυτών βασιζόταν στην διαχείριση των γεών και στην διατροφική επιστημιστική ε, αυτάρκεια. Απέχει πόρο από τα σημερινά, αυτά που συζητήσαμε το 2014-2020 στη νέα προγραμματική περίοδο. Σήμερα ε, δεν ανανεώνεται η οικονομική δραστηριότητα στις υπαίθριες περιφέρειες και πραγματικά απέχει επίσης πάρα πολύ πραγματικότητα και από αυτά που η ε, έκθεση ε, παρουσιάζει. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις χαμένες εκμεταλλεύσεις, ε, τις χαμένες γεωργικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία προοπτική στην έκθεση αυτή για τη γεωργία και οι υπαίθριες περιοχές όλο και περισσότερο γίνονται ε, ζώνες δεύτερης κατηγορίας ε, με πληθυσμό που γυράσκει, που, ε, την ήπειθρο που αποψηλώνεται και τώρα ακούμε ότι θα πάνε να εγκαταστήσουν εκεί μετανάστες. Λες και έτσι θα ξαναγεννηθεί η ύπεθρος. Στη Γαλλία βλέπουμε υπάρχει όλο και περισσότερη πελατειακή σχέση μεταξύ της περιφερειακής διοίκησης και κάποιων ε, φορέων της γεωργίας, γιατί αποδυναμώνεται η κεντρική διοίκηση και περνάει στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση. Αυτό για μας είναι αντίθετο με την αρχική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, παρακάπτεται η κεντρική εξουσία, ε, επικοινωνούν απευθείας με την τοπική αυτοδιοίκηση οι Αυτό είναι λάθος και στρατηγικό σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Και δεν ασχολούμαστε με το βασικό και μοιραίο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία που είναι η απελευθέρωση των αγορών. Ευχαριστώ. Ε. Μάλιστα, ναι. Αλλά το συζητάμε αυτό φυσικά στις ε, επιτροπές μας. Ο κύριος Μπούλερ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, παρουσίαση της, ε, του σχεδίου και θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στο ψητό. Στο θέμα της υπέτρου. Τον τελευταίο καιρό όλο και πιο πολύ επικεντρωνόμαστε στην αντίθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και μάλιστα αυτό το κάνουν ιδιαίτερως κάποιοι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Και νομίζω ότι για να είμαστε σωστοί όταν μιλάμε για χρηματοδότηση μεταξύ των χωρών της Ανατολής και της Δύσης, θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πραγματικά ακριβείς. Να μιλήσω για τη χώρα μου, τη Ρουμανία. 92% των κεφαλαίων που επενδύονται στη Ρουμανία είναι αλλοδαπά κεφάλαια. Και αυτές οι επενδύσεις γίνονται με τοπικούς πόρους. Αλλά 92% προέρχεται από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, στο θέμα και στον τομέα των αυτοκινούμενων οχημάτων, τα τρακτέρ. Ε. Και το ίδιο σημαίνει και σε άλλους τομείς. Παρόμοια κατάσταση. Πιστεύετε ότι είναι κακό ε, των να των επενδύσει στι ανατολικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι κάθε ευρώ το οποίο δαπανάται, επενδύεται στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, έχει διπλάσια άξια τελικά και έχει διπλάσια πόσο αποφέρει στους επενδυτές. Άρα θα πρέπει να μιλάμε και για το κέρδος, όχι μόνο για τις επενδύσεις και τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που επενδύονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ύπεθρο συγκεκριμένα, Φυσικά και όλοι θέλουμε να ενδυναμώσουμε τον τομέα της υπέτρου, προκειμένου να καταστεί ελκυστικός και προκειμένου να σταματήσει και η εγκατάλειψη της υπέτρου. Και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο θέμα, λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα, το ότι εγκαταλείπεται η υπεθρώση σταδιακά. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια διπλή αξιοποίηση των ταμείων αυτών για να καταπολεμηθεί η εγκαταλείψη τη υπαίθρου σε ό,τι αφορά τι υποδομέ, ε, την εκπαίδευση, το διαδίκτυο ε, και όλε αυτέ οι υποδομές οι οποίε τελικά έχουν ω αποτέλεσμα να υπάρχει και μεγαλύτερη θέση, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε βιώσιμε λύσει και για το μέλλον προκειμένου ακριβώ να υπάρξει ένα μέλλον για όσου ζουν στην υπαιθρο, κλείνοντα δύο παρατηρήσει, επιτρέψτε μου. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την υπερβολική γραφειοκρατία, να σας πω ότι συναντήθηκα με έναν ε, δήμαρχο από τη Ρουμανία, με ε, ότι συναντήθηκα λοιπόν με διάφορους δημάρχους στη Ρουμανία και μου ανέφεραν τέτοια θέματα γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία προκειμένου να μπορέσουμε πραγματικά να αναδείξουμε το δυναμικό τη κάθε περιοχής, γιατί θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθεί καλύτερα ο τομέας της υπαίθρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο ε, ακούγοντας διάφορες λύσεις, γιατί πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ε, θα ήθελα πάντα ε, καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ντανσίλα για ε, την εργασία της. Έχει κάνει και πολύ καλές προτάσεις. Δέκα χρόνια ήμουν, ε, δεκατών δηλαδή, όταν ε, είδα να υπογράφεται η συνθήκη της Ρώμης και έχω ζήσει όλη την εξέλιξη. Η Γερμανία ήταν μαζί ε, από τους πρώτους τα ιδρυτικά μέλη και τότε ήταν από τις φτωχότερε χώρες μετά τον πόλεμο και σήμερα είμαστε από τις πλουσιότερες. Ε, η εκλογική μου περιφέρεια έχει 1,7% ανεργία. Είναι δεύτερη ε, στη Γερμανία σε απασχόληση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματά της βοήθησαν πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Ήταν μια ε, καθυστερημένη περιφέρεια που αναπτύχθηκε και εκεί έχουν ευθύνη και τα κρατη τα προγράμματα που προσφέρονται από τις Βρυξέλλες θα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά και αυτό είναι ευθυνή και των κρατών μελών και στην Ήπεθρο. Εάν σήμερα στην Ήπεθρο δημιουργείται μια βιομηχανική, βιοτεχνική ζώνη και δεν υπάρχει ευρυζωνικότητα και γρήγορο διαδίκτυο, ποιο θα πάει να εγκατασταθεί. Και επειδή θα του πει ότι φτιάχνω μια βιομηχανική βιοτεχνική ζώνη, χρειάζονται επενδύσει κρατικέ. Αυτό που με έχει φέρει σε κάποια απόγνωση, γιατί είμαι εδώ πάνω από 12 χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για απλούστευση, για μείωση της γραφειοκρατίας κτλ. Τώρα σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πια για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγμα πραγματικά είναι αφόρητο όλο και περισσότερες ρυθμίσεις, διατάξεις, κανόνες. Δεν ξέρω, χρειάζεται έκτακτη επιτροπή για να ασχολείται με αυτό το θέμα επιτέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φτιαχτούν τα προγράμματα έτσι ώστε και άνθρωποι, ε, αγρότες, μικροί και όχι εταιρείε, ε, βιοτέχνες, ε, τεχνίτες, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι προηγουμένως Έχουμε άξια διοίκηση, αλλά έχουμε και πάρα πολύ σχολαστική διοίκηση και πάρα πολύ ε, συστηματική. Στη δική μου την περιφέρεια, το κρατήδιο της Βαβαρίας, δεν μας φτάνουν τα χρήματα από το δεύτερο πυλώνα. Έχουν απορροφηθεί και θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμόζονται και καμιά φορά άμα θέλετε να ανταλλάξουμε και εμπειρίες ε, για να μπορούν να εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά τα προγράμματα. Υπάρχει δυνατότητα. Και κατά τα άλλα θέλω να πω ότι και για τους νέους θα πρέπει να προσφέρουμε μαθήματα γλωσσών. Διάβασα πρόσφατα ε, ότι στην περιοχή μου υπάρχουν 500 ε, θέσεις άδειες μαθητείας. Και ακούω ότι έχουμε ε, νέους που ε, είναι άνεργοι 50% ενεργεία σε κάποιες χώρες. Όταν ήμουν εγώ μικρός ερχόντουσαν πολλοί Ισπανοί, Ιταλοί και Πορτογάλοι στη Βαβαρία. Γιατί δεν έρχονται να μάθουν μια τέχνη και ένα επάγγελμα. Πριν από 50 χρόνια ήταν πιο ευέλικτη. Σήμερα όχι, να το πούμε και αυτό. Γιατί έχουμε 500 θέσεις μαθητείας και νες που μπορεί ο άλλος να έρθει να μάθει ένα επάγγελμα, μια τέχνη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και εκεί μεγαλύτερη ευελιξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, την εισηγήτρια και πιστεύω ότι από κοινού θα το φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για την γνωμοδότησή της. Και θα ήταν καλό να την ενισχύσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμητικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της γεωργίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Πολύ σωστά μας υπενθυμίσει ο συνάδελφος ο Προλήσης ότι όλα ένα, μία θέση απασχόλησης στη γεωργία ανοίγει 7 επιπλέον θέσεις απασχόληση σε άλλους τομείς. Είναι σημαντικό λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα. Επίσης, πολλοί συνάδελφοι επισήμαναν τις περίπλοκες διαδικασίες και τις πολλές διατυπώσεις που ισχύουν και την ε, δύσκολη προσπέλαση σε δημοσιονομικά μέσα, κυρίως για τους ε, μικρούς και μεσαίους γεωργούς και τις μικρομεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να συμβάλλουμε με τη γνωμοδότησή μας ώστε να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί στην Κροατία Νιώθουμε την ανάγκη για απλούστευση της γραφειοκρατίας και για ταχύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στα κοινωτικά κονδύλια. Αυτό θα ανακουφίσει ιδιαίτερα τους Γιώργους και με βάση τις ε, τελευταίες, ε, στοιχεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια, περίπου 150.000 ε, νέοι μορφωμένοι άνθρωποι μεταναστεύουν λόγω έλλειψης προπτικών από την Κροατία και τα χωριά μας ε, και η Πεθρός μας απεριμώνονται. Καλό θα ήταν λοιπόν με τα κοινοτικά κονδύλια να ενθαρρύνουμε αυτούς τους νέους, να τους εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε αυτά τα, τα κοινοτικά κονδύλια για να παραμείνουν στην Ήπεθρο, να παραμείνουν στα χωριά και να ενισχυθούν και οι υποδομές των χωριών για της Ήπεθρου. Ας μην ξεχνούμε ότι τα χωριά είναι οι θεματοφύλακες της εθνικής ταυτότητας. Γι' αυτό και πραγματικά αξίζουν τις αμέριστες υποστήριξης μας. Ευχαριστώ. κυρία Κάντεμπαχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω και να σας ε, ταλαιπωρήσω γιατί αυτά που μας είπε ο κύριος Δέσσε προκάλεσαν έτσι διάφορες εξάρσεις. Είμαι μέλος και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και στην Αυστρία, στο κρατήδιό μου. Ήμουν μέλος και της Επιτροπής ε, ε, Ελέγχου Προπολογισμών και θα ήθελα να σας πω το εξή ότι διάφορες εκθέσεις και αυτές που λαμβάνουμε εδώ και έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και οι εκθέσεις οι οποίες ε, λαμβάνουμε από τα ελεκτικά συνέδρια στα κρατη είναι πράγματα τα οποία παίρνουμε στα σοβαρά. Γιατί είναι σημαντικά τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτές και διαπιστώνουμε ότι αυτές οι εκθέσεις από τα ελεκτικά συνέδρια, από τις ειδικές επιτροπές, ε, πάντα συζητιούνται βεβαίως, αλλά δεν έχουν τον αντίστοιχο και τον απαραίτητο αντίκτυπο, αν θέλετε, στις εργασίες των αρμόδιων επιτροπών χρηματοδότησης. Και αυτό δυστυχώς ισχύει και στα κρατημέλη. Και αυτό που ουσιαστικά συζητάμε είναι το πώς θα κατανείμουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια κινούμαστε προς την κατεύθυνση της ε, λογικής και σωστής ε, δαπάνης. Αλλά εδώ να έχουμε υπόψη ε, ότι χρειάζεται και κάποιο έλεγχο. Φυσικά συμφωνώ με όσου είπαν ότι θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και θα πρέπει φυσικά να εστιαστούμε σε καλύτερου, περιορισμένου και αποτελεσματικού ελέγχου. Και νομίζω ότι με την ε, Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη έχουμε καταθέσει πολλέ σημαντικέ και χρήσιμε προτάσει για τα κρατή μέλη και για τι διάφορε ε, ομάδε που ασχολούνται τον τομέα αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτέ οι προτάσει. Γιατί το χειρότερο θα ήταν να πούμε τώρα, Α, κοιτάξτε, είναι τόσο περίπλοκο το να λάβει κανεί επιδοτήσει. Α τα απλοποιήσουμε όλα. Α αφήσουμε και του ελέγχου και τι έγινε. Υπάρχουν πάρα πολλέ σωστέ προτάσει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν νέε επιτροπέ, νέε ομάδε. Θα πρέπει να α, ε, κοιτάξουμε πιο επισταμένο σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Μία μικρή παρατήρηση να κάνω. Σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ λυπάμαι που πιστεύουν κάποιοι ότι η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη είναι πολιτική κατανομής χρημάτων. Λες και αυτό είναι το επίκεντρο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ πιστεύω ότι περιλαμβάνει πολύ παραπάνω στοιχεία. Φυσικά περιλαμβάνει και αυτό το πώς ε, κατανείμονται οι πόροι, αλλά η πολιτική δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την ανάθεση πόρων, τη διανομή των πόρων. Δεν είμαστε μια επιτροπή διανομής. Δεν μπορούμε να το εξισώσουμε αυτό με την γενικότερη πολιτική αγροτικής ανάπτυξη. Εγώ έχω άλλη αντίληψη για την πολιτική ανάπτυξη. Στη συζήτηση αυτή θα πρέπει να προσέξουμε λίγο. Να μην παραφορτώσουμε τη ε, υπόθεση του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή να θέλουμε να χρηματοδοτούνται όλα από εκεί και υποχρηματοδοτείται και σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση είναι. Για το πρόγραμμα για την ενίσχυση των επενδύσεων θα πρέπει να ρωτήσουμε αν μπορούν να απορροφηθούν τα χρήματα. Τι γίνεται, ας πούμε, καταργήθηκαν γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Ε, δημιουργούνται νέες εκτροφές, νέοι στάβλοι, μετά δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το γάλα. Τι γίνεται, και όλα αυτά ήταν και χρήματα από το δεύτερο πυλώνα. Θα πρέπει και αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη. Εξού και είναι σημαντικό βεβαίω να έχουμε προγράμματα στο δεύτερο πυλώνα βεβαίως για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και εγώ απορρίπτω και αποκρούω αυτά που ακούμε από τη δεξιά και την ακροδεξιά για τη μετανάστευση που το κάνει τέτοιο θέμα. Φυσικά θα πρέπει οι άνθρωποι να ενταχθούν και στην Ήπεθρο. Πού αλλού θα τους βάλουμε. Εκεί που δημιουργούνται θέσεις εργασίας θα πρέπει να μπορούν να απασχολούνται και οι πρόσφυγες και να έχουν ε, καμιά προοπτική για το μέλλον τους. Και τώρα να δημιουργούμε εντυπώσει κατά των προσφύγων που στο κάτω-κάτω χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους για να ενταχθούν στην κοινωνία, το θεωρώ παράλογο να το συζητούμε εδώ μέσα. Και μια πρόταση προς τον κύριο Ντες. Αν υποχρηματοδοτούνται τα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα και ε, στη Βαβαρία και αλλού, υπάρχει δυνατότητα μεταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Και περιμένουμε μεγάλη περιέργεια να δω τι θα πούνε οι Τσέσου και οι Τσέντεου χριστιανοδημοκράτες ε, στη Γερμανία. Γιατί αν υποχρηματοδοτούνται, βάλτε τα λεφτά από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Μήπως γίνεται καλύτερη πολιτική έτσι από το καταποκοπή να μοιράζουμε λεφτά από τον πρώτο πυλώνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος να ξαναζήτησε το λόγο. Μία παρατήρηση να κάνω, Πρόεδρε τα χρήματα του πρώτου πυλώνα δεν τα πήγαμε στο δεύτερο πυλώνα. Η Βαβαρία αποφάσισε σε διαδικασία ελέγχου να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετη πορεία στον προπολογισμό. Δεν αφαιρούνται από κάπου αλλού αυτά τα χρήματα δηλαδή. Δεν έγινε απλά μια μετακίνηση. Είναι επιπρόσθετη πόρη για την χρηματοδότηση των στόχων αυτών. Ναι, είχατε από πού να τα πάρετε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπούσα από τη Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω απλά ότι η έκθεση αυτή, η ανακοίνωση αυτή ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Άρα, ουσιαστικά παρουσιάζει τα όσα είχαν εντοπιστεί και όσα είχαν συμφωνηθεί ε, μεταξύ των κρατών μελών και τα διάφορα προγράμματα και ασφαλώς για αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο συνεχίζει τη συζήτηση περαιτέρω για το τι ε, θα πρέπει να γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής μας και σε ό,τι αφορά την ε, διανομή των πόρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση της συγκεκριτρίας, την οποία και καλωσορίζω, χαιρετίζουμε το νέο στοιχείο της, ε, των τοπικών ε, ε, ομάδων δράσης. Το καλωσορίζουμε. Είναι πραγματικά μια καινοτομία αυτή στην νομοθεσία. Πολύ ευπρόσδεκτο και ελπίζουμε πραγματικά να το χρησιμοποιήσουν και να το εκτιμήσουν τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο το οποίο συγκρατώ από τη σημερινή συζήτηση είναι το ότι θα πρέπει να απλοποιήσουμε την πολιτική μας και θα πρέπει να καταβάλουμε πάσα προσπάθεια προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητή, πιο διαφανής, να αποφεύγονται οι έλεγχοι, να αποφεύγονται οι ατασταλίες. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση που ζητά από τους δικαιούχους να συμβάλλουν προ την κατεύθυνση τη απλοποίηση. Να δούμε τι πιστεύουν δηλαδή και οι ίδιοι δικαιούχοι, οι ίδιοι αγρότε. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα προκειμένου να βελτιώσουμε την πολιτική αυτή για το μέλλον. Και αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα έχει... Θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια πορίσματα τα οποία θα ληφθούν υπόψη και για τι μελλοντικέ συζητήσει τη αναπτυξιακή πολιτική. Και φυσικά να μειωθεί η γραφειοκρατία. Θέλουμε ασφαλώς να παραμείνει και ένα στοιχείο ευελιξία. να είμαστε ανοιχτοί και προς νέους ε, κανόνες και ενδεχομένω πάντα υπάρχει το προφανές ε, ζήτημα του τι θα κάνουμε, θα ε, προτιμήσουμε νέους κανόνες ή θα απλοποιήσουμε τους παλιούς κανόνες. Πάντα αυτό μας απασχολεί. Και μια άλλη παρατηρήση, επιτρέψτε μου. Για αυτά που είπε κάποιος βουλευτές, ότι εκβιάζουμε τα κρατημέλη. Δεν εκβιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κρατημέλη. Όχι, εφαρμόζουμε απλά την νομοθεσία την οποία μεταξύ άλλων έχει υπερψηφίσει και το Κοινοβούλιο. Το άρθρο 24, για παράδειγμα, τη κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Ε, απλά σεβόμαστε λοιπόν την νομοθεσία η οποία ήδη υφίσταται. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ε, εκδοχή εκβιασμού. Σας ευχαριστώ και τώρα η συγκεκριά μας. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας ε, και όλες τις διευκρινήσεις που κάνατε με τις παρατηρήσεις σας. Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε με την πείρα μας και να καταρτήσουμε τροπολογίες προκειμένου να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση. Έτσι θα την εμπλωτίσουμε και θα την κάνουμε πιο πλήρη και μεστή, χάρη και στις τροπολογίες που θα υποβάλλουν οι συνάδελφοι και με τις οποίες θα συμπληρώσουν μερικά σημεία που ίσως μου διέφυγαν. Σας ευχαριστώ και περιμένω με αδημονία τις τροπολογίες σας. Μάλιστα. Έχουμε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου ε, στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και επίση να υπενθυμίσω ότι η υπεθρός δεν περιορίζεται στη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική αφορά την γεωργία. Το, ο δεύτερος πυλώνας αποτελεί ένα τμήμα της γεωργικής πολιτικής, αλλά η υπεθρο έχει δικαίωμα και είναι και επιλέξιμη και για τα κονδύλια της συνοχής, για να εξασφαλιστεί μια εδαφική συνοχή. Οπότε η μπορεί να υποφελείται και από ε, το Ταμείο το Κοινωνικό και το Ταμείο Συνοχής για να απτυχθεί. Και υπάρχουν κάποιες πτυχές που συνδέονται με τη γεωργία. Έτσι θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε το όλο οποίο Η γεωργία είναι ένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν το τοπίο της υπαίθρου. Σημαντικό μεν, αλλά δεν είναι το μόνο. Η υπεθρός είναι ευρύτερη, είναι δεν με τη γεωργία και καλύπτει και άλλους τομείς. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη γιατί έχουμε και τα ταμεία συνοχής που μπορούν να ενισχύσουν την υπεθρό. Αυτά για να αποφύγουμε κακές αποφάσεις. Ολοκληρώνουμε με την δημόσια συνεδρίαση, το δημόσιο τμήμα της συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε στις 3 και θα περάσουμε τώρα στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε παρακαλώ τους συντονιστές ε, να είναι στην αίθουσα στις 11 για να αρχίσουμε λίγο νωρίτερα τη συνεδρίαση. Και επίσης ε, θα ήθελα να έχουμε την επιβεβαίωση ε, από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, γιατί ίσως κάποιοι συντονιστές έρθουν στις 11 και 4 που αρχικά ήταν η προβλεπόμενη ώρα. Παρακαλώ, οι βοηθοί και οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων να φροντίσουν ώστε να είναι παρόντες στην αίθουσα για την έναρξη της συνεδρίας των συντονιστών στις 11 οι συντονιστές. Αυτά σας ευχαριστώ.